Εάν το κάνετε αυτό θα μας έχετε στο πλευρό σας για να αλλάξει επιτέλους ο κανονισμός. Κύριε Μαν, αντιλαμβάνομαι την απογοήτευσή σας και εμένα δεν μου αρέσει να μην μπορώ να δίνω στους συναδέλφους τον λόγο για τόσο σημαντικά ζητήματα, αλλά επίσης σωστά λέτε πως απαιτείται να αλλάξει ο κανονισμός του Κοινοβουλίου γι' αυτό. Οπότε, ειδού. Και αυτό το οποίο θα προσέθετα είναι πως εάν όλοι οι συνάδελφοι σέβονταν το χρόνο τους θα μπορούσαμε να ακούσουμε περισσότερους συναδέλφους. Φοβάμαι πως αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε θα περάσουμε τώρα στη ψηφοφορία. Ούτως ή άλλως τα σχόλιά σας έχουν σημειωθεί. Έχουμε λοιπόν τα 7 ψηφίσματα για την θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν και νομίζω πως ο κύριος Πόσελτ θέλει να καταθέσει μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 13. Κύριε Πρόεδρε, έχουν λειτουργήσει πάρα πολύ καλά οι συνάδελφοι. Έχουμε φτιάξει ένα θαυμάσιο ψήφισμα μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων. Αλλά έχει καταλήξει στην παράγραφο 13 ένα κείμενο το οποίο είναι λιγάκι συγκεχημένο. Γι' αυτό εμεί θέλουμε να προτείνουμε μια νέα διατύπωση, εκφράσει την ανησυχία του για την δυνατή ε, αρνητική αντιμετώπιση της εκστρατείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπογραμμίζοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η νέα διαδικασία θα πρέπει να εγκριθεί από την Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ κύριε Πόσελτ. Υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι, δεν φαίνεται. Μπορούμε να την θέσουμε σε ψηφοφορία λοιπόν. ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική ε, γνώμη Β σε δύο τμήματα ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές θα ήθελα να έχουμε λοιπόν ένα ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της αιτιολογικής σκέψης Β, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Β, λατινικό 5, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Το κοινό ψήφισμα λοιπόν ως σύνολο ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Ακολουθεί, ακολουθούν τα έξι ψηφίσματα για την Ταϊλάνδη. Έχουμε τροπολογία 4 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 6 παρακαλώ Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη α σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι κατά, αποχές, δεκτό δεύτερο τμήμα, ψήφι κατά, αποχές, δεκτό. Τροπολογία 2, ψήφι κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Το κοινό ψήφισμα <clears throat> ως έχει τροποποιηθεί ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτό. Περνάμε στα 7 ψηφίσματα για τη Βυρμανία. Χωρίς τροπολογίες θέτω το, τα ψηφίσματα, το κοινό ψήφισμα σε ψηφοφορία μονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Γίνεται δεκτό το κοινό ψήφισμα για τη Βερμανία. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συντάκτες των ψηφισμάτων τα πρακτικά της συνεδρίασής μα θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο για την έγκρισή του στην έναρξη της επόμενης συνόδου. Εάν δεν έχετε καμία αντίρρηση, θα διαβιβάσω τα ψηφίσματα τα οποία εγκριθήκαν στους φορείς που αναφέρονται στα οικία ψήφισμα. Η, ε,